κατά αποχές απορρίπτεται Ένα. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Δώδεκα. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Δύο. υπέρ κατά αποχές check two. Επαλήθευση για τη δύο, παρακαλώ Πέρας φοβορίας εγκρίνεται. Ε, τρία και δέκα μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31 παράγραφος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 51 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 54 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 59. Υπέρ. I'm sorry. Ναι, τροπολογία 5 στην παράγραφο 59, με συγχωρείτε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 64 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Check. Check. Paragraph 75. Παράγραφος 75, ηλεκτρονική επαλήθευση, παρακαλώ. Did I do paragraph 75? Yes, you did. No, no, that was before. because you always have to, you very often have a Okay, my, my, my mistake, my mistake. Let's go back. Εγώ έκανα λάθος. Ε, γυρνούμε προς τα πίσω τώρα. Επιστρέφουμε στην τροπολογία 6, παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 89 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 90. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος τροπολογία 9. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 108. Σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Check. 7. Την 7 έλεγχος παρακαλώ. Ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας απορρίπτεται τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Α, ε, αιτιολογική σκέψη F σε δύο μέρη πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τέλικη ψήφος ποιοι είναι υπέρ ποιοι είναι κατά αποχές Εγκρίνεται. Ευχαριστώ κύριε Σάλτη. Ακολουθούν τώρα οι επεξηγήσεις ψήφου.